el señor presidente. Buenos días, colegas. Πολύ καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Έχω μία ανακοίνωση. Ζητήθηκε από τον κύριο Πυρίλο διαδικαστικό. Ευχαριστώ κύριε